Uh, Έχω ενημερωθεί πως η κυρία Κοράτσα Μπίλτα έχει διαδικαστικό να ζητήσει. Παρακαλώ ας ακούσουμε τη συνάδελφο. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να εγείρω ένα ζήτημα πάτης ως προς την ψηφοφορία της κυρίας Λεπέν. Αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε να συνεχίσω. Έχω παρακαλώ, παρακαλώ τους αδέλφους, λέει ο Πρόεδρος, τουλάχιστον να δείξουν αρκετό σεβασμό ώστε να ακούσουν τι έχει να πει η κυρία Ράτσα Μπίλτ. Τον, Οκτώβριο, λοιπόν, τον Νοέμβριο λοιπόν έγινε ένα ζήτημα και είχατε πει ότι θα, ε, θα αναπτύξετε μια έρευνα της υπόθεσης αυτής. Περιμένουμε ύστερα από τόσους μήνες αποτελέσματα. Ο κύριος Μάρσελ Ντεγκράφ, συμπροεδρεύων της ομάδας των Ευρωπαϊκών Εθνών και της Ελευθερίας, έχει καταδικαστεί για εξαπάτηση ως προς την ψηφοφορία σε πρωτοβουλία πολιτών, αλλά για τον κύριο Μπέ δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση για την ψηφοφορία τη σχετική με τις εκπομπές καυσαερίων και την, ε, τα, αυτά οχήματα. Έχετε κάτι να μας πείτε για τον κύριο Μπέ και την ε, απάτη στην ψηφοφορία κύριε Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος. Οφείλω να σας ενημερώσω πως επιφορτίστηκα από τον Πρόεδρο ξεκινώντας να προβώ στην ανακοίνωση την οποία θα σας αναγνώσω μέσω μετά και η οποία σχετίζεται με το συγκεκριμένο περιστατικό. Η κυρία Λεπέν όμως ζήτησε το λόγο και την παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κυρία Καρατσαμπίλτ φαίνεται να έχει αναπτύξει μια μονομανία ως προς το πρόσωπό μου και την ευχαριστώ. Την ενημερώνω πάντως ότι αντίθετος προς τις ψευδείς και δυσφημιστικές ε, κατηγορίες που αναπτύσσει βάρος μου, έχω αθωθεί απολύτως την υπόθεση αυτή. Ο πρόεδρος. Όπως είπα, πρόκειται για τα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Θα διαβάσω λοιπόν το κείμενο της ανακοίνωσης που μου δόθηκε και μου ζητήθηκε να παρουσιάσω εκ μέρους του Πρόεδρου. Αρχίζω λοιπόν την παράθεση. Όπως ασφαλώς ενθυμίστε, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια της 28 Οκτωβρίου του 2015, ο Πρόεδρος εκλήθη από την κυρία Κοράτσα Μπίλτ να επαληθεύσει τις συνθήκες υπό τις οποίες η ε, μηχανή για την ψηφοφορία της κυρίας Λεπέν χρησιμοποιούνταν τη απουσία της στις 17 Δεκεμβρίου του 2015. Το Κοινοβούλιο ενημερώθηκε για την απόφαση του Προέδρου να επιβάλει κύρωση στον κύριο Ντεγκράφ για την συμπεριφορά του κατά την εν λόγω ψηφοφορία, δηλαδή διότι χρησιμοποίησε τη μηχανή της κυρίας Λεπέν. Η κύρωση συνίστατο στην στέρηση του ενός ε, του ισοδυνάμου πέντε ημερών ημερησίας ζημίωση. Επίσης και ύστερα από ε, ακρόαση με αρκετούς βουλευτές και τον κύριο Μπέ Δις, ο κύριος ε, Πρόεδρος αποφάσισε να επιβάλλει αντίστοιχη κύρωση στον κύριο Μπέ για την συμπεριφορά του, δηλαδή τη χρήση αντίστοιχα του μηχανήματος για την ψηφοφορία της κυρίας Λεπέν. Η κύρωση θα είναι στέρηση ισοδυνάμου πέντε ημερών της ημερήσης αποζημίωσης. Έχει ενημερωθεί ο εν λόγω βουλευτής για την απόφαση του Προέδρου. Κύριε Μπέ. Κύριε Πρόεδρε, η παρέμβασή μου βασίζεται στα άρθρα 164 και 167 του εσωτερικού κανονισμού. Θα καταθέσω μία έφεση απέναντι σε αυτήν την απόφαση που δεν έχει καμία νομική βάση και καμία απόδειξη. Η απόφαση του Πρόεδρου σου δείχνει την ολοκληρωτική μορφή της διαχείρισης την οποία εφαρμόζει. Το έδειξε και την προηγούμενη Τρίτη μπροστά στον εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών. Οι κατηγορίες αυτές ε, είναι προϊόντα φαντασίας και μαρτυρίες οι οποίες δεν υπήρξαν ουσιαστικά ποτέ, δεν επαληθεύθησαν ποτέ και είναι και εναντίον του άρθρου 166 του εσωτερικού κανονισμού. Δεν οφείλω εγώ να αποδείξω την αθωότητά μου, θα πρέπει οι κατηγοροί μου να το αποδείξουν και οι τέσσερις από τους πέντε παραμένουν ανώνυμοι. Άλλωστε και ο ίδιος ο κύριος Σούλτς έχει ξεκινήσει για μια νέα ε, ημίσια ε, προεδρική εντολή και δεν θα υποκύψουμε ποτέ στα κραπίτσια των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ή άλλων. Καλώς. Σημειώνουμε την απόφασή σας να προσβάλετε την επιβολή κυρώσεων. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτζιτσε τώρα το λόγο. Πρόεδρε, πολύ σύντομα θα ήθελα να σημειώσω ότι πρόκειται για μια δημόσια διατύπωση mensonge, θα το πω στα γαλλικά, ψέμα, mensonge. Ο κύριος Μπέ ο ίδιος μου είπε ότι ψήφισε αντί για την κυρία Λεπέν. Πηγαίναμε με το αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο και έχω μάρτυρα την κυρία Φεντερικ Κρέης και αυτό δείχνει πως το Front National, το Εθνικό Μέτωπο, ε, νομίζει ότι μπορεί να έρεται άνω των κανόνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος. Κοιτάξτε, εγώ είχα να κάνω την, την ανακοίνωση για τον κύριο Μπέ και την ανακοίνωση της κύρωσης